Δεν ήταν και τόσο εντός θέματος, αλλά σας ευχαριστούμε. Please stay in είναι ο Κάρλος Κουέλιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε κύριε Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε Κίνγκ, οι ευρωεκλογέ στο Μαΐο, οι πολίτε θα πρέπει να επιλέξουν ποιον θέλουν ή να του εκπροσωπήσει το μέλλον. Και αυτή η επιλογή του θα πρέπει να είναι ελεύθερη. Δεν θα πρέπει να δώσουμε λαβή σε όποιον θέλει να καταστρέψει το ευρωπαϊκό όραμα. Υπάρχουν εξωτερικέ δυνάμει που θέλουν να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν συμμάχου εδώ μέσα. Και όπω είδαμε πρόσφατα, είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν όλα τα όπλα που έχουν στη διάθεσή τους, ιδιαίτερα τα ψηφιακά όπλα. Ε, γνωρίζουμε όμως αυτές τις απειλές. Ε, το 70% των πολιτών ανησυχούν για εκστρατείες παραπληροφόρηση. 77% ανησυχούν για, τα, για παραπημένα αποτελέσματα. Και ε, ε πολλοί κόσμος ακόμα ανησυχεί όσον αφορά τις δημόσιες παρεμβάσεις. Πρέπει λοιπόν να καλύψουμε τα εκλογικά θέματα και να θωρακιστούμε απέναντι σε οποιαδήποτε πληροφοριακή επίθεση. οι ψηφιακές πλατφόρμες ε, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να συνεργαστούν μαζί μας και να αποφύγουμε τα fake news, τις ψευδείς ειδήσει. Η ελευθερία, η δημοκρατία και κράτος δικαίου είναι οι αξίες μας, είναι η ταυτότητά μας, είναι η ταυτότητά μας που κάποιοι θέλουν να καταστρέψουν με νέα όπλα. Το να την υπερασπιστούμε δεν είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβουμε, είναι μια υποχρέωση στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος τώρα των σοσιαλιστών, ο κ. Φρόιντ. Να πω εξ ότι αυτό, δεν θα πρέπει να είναι κομματικό θέμα. Θα πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι στην αγώνα κατά των ψευδών ειδήσεων, της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας. Φοβούμαι όμως ότι αυτό είπε και ο κύριος Τέλιτσκα, ότι τα κράτη-μέλη δεν γνωρίζουν αυτό το θέμα και δεν προσέχουν αρκετά τις εντάσεις που προκύπτουν από αυτό. Δεν θα συνεχίσω στα γερμανικά, κύριε Κίνγκ. Το διαδικτυακό περιβάλλον ε, που έχει κατασταθεί τα τελευταία χρόνια φέρνει πολλές θετικές αλλαγές. Όμως, δίνει όπλα και στους ε, αντιπάλους της δημοκρατίας ε, και του κράτους δικαίου. Το επέδειξε το Brexit και η εκλογή του Τραμπ ο επηρεασμός ε, της κοινή γνώμης αυξάνεται και είναι τόσο μεγάλος ο βαθμός που οι δημοκρατικές εκλογές μπορεί πραγματικά να επηρεαστούν. Οι εξελίξεις αυτές θα υπάρξουν και στις επικείμενες ε, ευρωεκλογές. Θα είναι πρόβλημα. Εάν μια ψευδής είδηση αρχίσει να κυκλοφορεί, τότε θέλουμε χρόνο μέχρι να την αντικρούσουμε. Επιπλέον, έχουμε την τεχνική πρόοδο. Και εδώ δεν θα πρέπει να βραδιπορούμε έναντι των τεχνικών εξελίξεων. Γιατί πέρα από τα κλασικά κανάλια κοινωνική δικτύωση, Facebook, Instagram, Twitter, υπάρχει και το WhatsApp, το οποίο παίζει έναν ε, αμφισβητούμενο ρόλο. Και η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά δυνατό να διαδίδεται προπαγάνδα και ψεύτικε ειδήσει σε τεράστιες διαστάσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εγγυηθεί την νομιμοποίηση των ευρωεκλογών. Τότε πρέπει να εντοπίζει αυτά τα φαινόμενα τάχιστα και να τα παρεμποδίζει. Χρειαζόμαστε μία καλή στρατηγική για να αντιμετωπίζουμε την διάδοση ψευδών, μισοαληθιών και την προσπάθεια περιορισμού της διαμόρφωσης της κοινή γνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Υπάρχει μία κάρτα για σας. Τη δέχεστε. Ωραία. Κύριε Ρούμπιχ, ποια είναι η ερώτησή σας. Ναι. ναι. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Φρόιντ. Ω δημοσιογράφο ε, αναγνωρίζει καλά τα θέματα αυτά. Τη βδομάδα αυτή είχαμε το θέμα για την ε, ασφάλεια. και θα πρέπει λοιπόν και τα 28 κράτη-μέλη να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις γι' αυτό. Υπάρχει και το ΣΤΟΑ που έχει κάνει τέσσερις μελέτες για την κυβερνοασφάλεια. Και έχουμε δημιουργήσει και ένα μπόλο ε, για τα μέσα και την επιστημονική εξέλιξη. Θεωρείτε ότι επαρκούν αυτά τα μέτρα ή θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Παρακαλώ απαντήστε, κύριε Φρόντ. Ποτέ, αγαπητέ ε, Ρούμπιχ, δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει κάνει τα πάντα αρκετά για να είναι αποτελεσματικός. Φοβάμαι ότι για την επιρροή στις ευρωεκλογέ ε, έχουμε καθυστερήσει. Πρέπει οπωσδήποτε να μας απασχολήσει ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Γιατί αλλιώς μπορεί να προκύψει μια κατάσταση όπως αυτή με την εκλογή του Τραμπ και το, την έκφαση του δημοψηφίσματος για το Brexit. Τζαμπάσκι, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σίγουρα η δημοκρατία μας είναι κάτι που πρέπει να το προστατεύουμε και να το διαφυλάτουμε. Πολλοί εκπρόσωποι εδώ μέσα φοβούνται ότι οι ευρωεκλογέ θα διαστραφούν μέσω της παρέμβασης ε, διαφόρων όπως η ακροδεξιά και άλλοι δεξιοί. Οι δυνάμεις αυτές θεωρούνται ανεδείς και στην ουσία τι μας λένε ότι εάν ένα από αυτά τα κόμματα τα πάει καλά στις εκλογές αυτό οφείλεται στην παρέμβαση ξένων παραγόντων. Ακούμε ότι παρεμβαίνουν ιδιαίτερα οι Ρώσοι που υποτίθεται βοήθησε την εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ. Ναι, αλλά η έκθεση Μίλλερ δεν ε, διαπίστωσε τίποτα τέτοιο. Αν θα σας αρέσουν τα αποτελέσματα των εκλογών, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αποτέλεσμα χειραγώγησης. Αυτό που λέτε ότι οι λαοί δεν μπορούν να αποφασίσουν ε, με λογικό τρόπο. Η κυρία Σχάκη. Τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών ε, διακυβεύονται μέσω της δυνατότητας ε, παρέμβασης ή ε, παραπλάνησης των πολιτών για να ψηφίσουν κάτι που ανεξάρτητα μπορεί να μην το ψήφιζαν. Και οι ψευδείς ειδήσει διαδίδονται στα μέσα όπως η πυρκαγιά. Πρέπει να επαγρυπνούμε και βλέπουμε τις ad hoc ε, προσπάθειες που, που υπόσχονται οι πλατφόρμες όπως ε, το YouTube, ε, το Facebook κλπ. Όμως θα πρέπει χωρίς, τις, χωρίς αλγορίθμους και χωρίς έρευνα δεν μπορούμε να πούμε στα σίγουρα ποιο είναι ο αντίκτυπο της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας στη δημοκρατία μας και αυτό είναι παράδεκτο. Πρέπει τώρα να δράσουμε. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Στέασης ε, έκανε ε, αγωγή κατά του Facebook γιατί ε, η πλατφόρμα αυτή έκανε διακρίσεις σύμφωνα με το Υπουργείο. Δηλαδή ότι δεν επιτρέπεται εκτός της πλατφόρμας, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται ούτε στις πλατφόρμες θα πρέπει να κάνουμε και ειδικέ δοκιμές για την τεχνολογία ε, της πληροφορίας. Δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο. Και τέλος θέλω να κάνω έκκληση σε όλους, σε όλα τα πολιτικά κόμματα της Ευρώπης, ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Καλώ τους συναδέλφους και τους ε, συνυποψήφιους για τις ευρωεκλογέ να υπογράψουν όλη τη δέσμευση στο, ε, για τις εκλογές στο electionpledge.eu ε, γιατί πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Η Ευρώπη είναι τόσο ισχυρή όσο είναι ο πιο αδύναμος κρίκος μας και θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Τάραντα, ένα λεπτό. The integrity of electoral systems is must η προστασία των εκλογικών συστημάτων είναι ε, υποχρεωτική, αλλά επίσης σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε την ε, συνολική ακυρότητα των ευρωεκλογών και να εμποδίσουμε την ε, αθέμητη παραπληροφόρηση από οργανισμούς όπως η Cambridge Analytica και σχετική και παραπλήση. Τα όσα είπε η συνάδελφος Χάκη τώρα τα συμμερίζομαι, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι το Facebook είναι μια τόσο τεράστια εταιρεία και εμείς ως νομοθέτες θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι ώστε να την καταστήσουμε υπεύθυνη ε, γιατί έδωσε στοιχεία ε, ε, σε τρίτα μέρη, όπως η Cambridge Analytica που ανέφερα προηγουμένως. Ε, ε, ε, από τη στιγμή που έχουν δοθεί τα, τα, δεδομένα δεν υπάρχει τρόπος να τα ξαναπεριορίσεις γιατί αυτά μπορούν να αντιγραφούν και να μοιραστούν παόριστον. Θα πρέπει λοιπόν το Facebook να, να προσέχει τα στοιχεία των χρηστών του ή διαφορετικά να απαγορευτεί ή ότι άλλο αποφασίσουμε εμείς. Σας ευχαριστώ και βγείτε από το facebook, θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Εγώ το έκανα και είμαι πολύ ευτυχής. Ευχαριστώ. Κύριε Τάραντ, υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας, τη δέχεστε? Την κυρία Γκραπίνη. Η ερώτησή σας παρακαλώ. Αξιότιμε συνάδελφε, είπατε μεταξύ άλλων και συμφωνώ πως υπήρξε χειραγώγηση μέσω πλατφορμών όμως από την άλλη πλευρά λέτε ότι δεν σας αρέσει το Facebook. Όμως πρέπει κανείς να στηρίξει ε, ε, την ψηφιοποίηση. Τι να κάνουμε λοιπόν εάν το Facebook πέρα από τις δικές μας προειδοποιήσεις ε, διατηρεί τους ψεύτικους λογαριασμούς όταν κάνει, μπορεί ας πούμε, να μπλοκάρεις κάποιον και μετά εμφανίζεται εκ νέου. Πώς μπορούμε να εξελίξουμε αυτές τις απειλές, ειδικά τώρα πριν τις ευρωεκλογέ. Κύριε Τάραντα, ποια είναι η απάντησή σας. Μακάρι να ήμουν τόσο έξυπνος για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Συμφωνώ με το όσο η Μαράια, ότι δεν επιτρέπεται ε, στην κανονική ζωή, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται ούτε και στην επιγραμμική ζωή. Γιατί εγώ έκλεισα το λογαριασμό μου στο Facebook και τα περισσότερα σχόλια ήταν «θα σε σκοτώσω». Ε, άτιμε. Πώς... Το έσβησα λοιπόν και εγώ τελείω το λογαριασμό και εισήχασα. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναπτυχθεί η ψηφιοποίηση, αλλά πρέπει να ελέγχεται, να είναι σε ανθρώπινες διαστάσεις, να είναι σε ανθρώπινος χώρος και όχι ένας χώρος απάνθρωπος και βίαιος. Ε, ε. Ο κύριος Βρετών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι ευρωεκλογέ θα πρέπει να είναι ελεύθερε και ε, ε, δίκαιες. Ε, είμαι υπέρ λοιπόν ενό εγγράφου που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση εξτατιών παραπληροφόρησης. Επίσης θα πρέπει να χαιρετήσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τι εκλογέ, χωρί να θυγεί η κυριαρχία του. Ωστόσο, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των θεσμών ενάντια στη τάση να, να, να δώσουν συγκεκριμένα φόρματ στην πληροφορία. Τα εθνικά κόμματα έχουν το δικαίωμα να επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προτείνουν την αντικατάστασή της από την Ευρώπη των Εθνών. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, εκτός και αν θέλουμε να βλάψουμε την πολιτική ελευθερία, ότι αυτή είναι στην καρδιά των ευρωπαϊκών δημοκρατιών. Κύριος Ράντεφ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πέτροπε, κυρίες και κύριοι, πρόσφατα άλλαξε σημαντικά το πλαίσιο και είδαμε αρκετές επιθέσεις από κυβερνητικούς και μη παράγοντες ε, από, την, ε, από το ιστορικό και το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, πει, κατα, αποτελούν σημαντική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες αποκομπήσουν την εντύπωση ότι είναι ευάλωτες οι δημοκρατίες όταν μπορούν να πληγούν έτσι εύκολα. Έτσι λοιπόν τα πιο το πιο δημοκρατικό ευρωπαϊκό όργανο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να ανανεωθεί με εκλογές που θα πρέπει να μην σεμεριμνήσουμε να είναι ανώθευτες και να μην αφήνουν καμία σκιά νομοποίηση σε σχέση με μια κυβερνοεπίθεση. Εδώ πρέπει να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με κυβερνοεπιθέσεις αλλά και συνεργασία μεταξύ των αρχών των αρμόδιων για την αντιμετώπιση του κινδύνου των απειλών από τον κυβερνοχώρο και γι' αυτό θεωρώ ευπρόσδεκτη την προσπάθεια για συντονισμό από τις Εθνικές Αρχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις προσωμιώσεις που θα πρέπει να επαναληφθούν και σε επίπεδο κράτους μέλους, ώστε κάθε κράτος να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει ενδεχόμενε κυβερνοεπιθέσεις εν των ευρωεκλογών. Και θέλω να καταστώ πολύ το σαφές ε, το ότι εάν τυχόν αμφισβητηθεί έστω και σε ένα κράτος μόνο η εκλογική διαδικασία, κινδυνεύει ολόκληρο το ευρωπαϊκό σύστημα εκλογικών αναμετρήσεων. Πράγμα το οποίο θα ικανοποιήσει οπωσδήποτε αυτού που θέλουν να μα κάνουν κακό και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κόφοντ, για ε, ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συζητούμε σήμερα εμεί ω όργανο νομοποιημένο και προσωπούν του Ευρωπαίου πολίτε, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να προχωρήσουμε στι ευρωεκλογέ χωρί να κινδυνεύουμε από οποιαδήποτε επίθεση προερχόμενη από τον κυβερνοχώρο, αλλά και οποιαδήποτε ανάμειξη σε ανώθευτε και γνήσιε ευρωεκλογέ. Α μην είμαστε όμω αφελεί. Ήδη έχουμε δει απειλέ και θα δούμε και άλλε απειλέ ει βάρο τη διαδικασία των ευρωεκλογών. Έτσι λοιπόν πρέπει οι πλατφόρμε να είναι απολύτω διαφανεί, να λογοδοτούν, να ακολουθούν την νομοθεσία με και αυτό σημαίνει βέβαια ότι η κοινωνία και η διαγραμμική πρέπει να είναι απολύτω διαφανής. Δημοκρατία βέβαια σημαίνει και ταυτόχρονα τρόπο ζωής νοοτροπία δημοκρατική. Πρέπει όλα τα κόμματα να, να υποστηρίξουμε την αλήθεια, να ταχθούμε στην αλήθεια και να καταπολεμήσουμε όλους αυτούς που μετερχόμενοι το ψέμα προσπαθούν να πλήξουν τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κάριμ. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το το δίχτυ έχει υφανθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει μπει κανένα κράτος αλόβητο. Υπάρχουν πολιτικοί φορείς ήδη με ψόγο και με στίγματα πάνω τους που κάθονται ακόμα και στα δικά μας έδρανα. Στη δική σας τη χώρα, τη δική μας πατρίδα κύριε Επίτροπε, το Ηνωμένο Βασίλειο, κάποιοι ε, δημοσιογράφοι αφέθηκαν μόνοι τους όπως ο Βάλτερ, ο Μπράιεν να ε, ξετρυπώσουν το τέρας. Το Brexit προέκυψε μέσα από ε, τον Collins, ε, επικεφαλής της Επιτροπής Σουόρτ ε, και ψηφιακών δεδομένων μέσα από το Facebook. Και να που τώρα αναδεικνύεται και ένα κόμμα Brexit που μπορεί να χρηματοδοτείται με ποσά μικρότερα των 500 λιρών χωρίς έλεγχο ποσά τα οποία εισραίουν ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Φαράς, πείτε μας από πού έρχονται τα χρήματα που σας χρηματοδοτούν το κόμμα. Ευχαριστώ πολύ. Φαρία, ένα λεπτό και τριάντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να αντισταθεί στις διεθνείς ε, ε, απειλές. Μετά από το σκάνδαλο όμως της Cambridge Analytica δεν μπορεί παρά να ε, αναγνωρίσει ότι επηρεάζουν οι πλατφόρμες Google, Facebook και λοιποί τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Και επίσης ε, υπάρχουν λαϊκιστικές δυνάμεις που θέλουν να παραλύσουν τις ευρωεκλογέ. Ο κίνδυνος ε, της επιρροής των επόμενων ευρωεκλογών από fake news και από παραπληροφόρηση είναι πολύ σημαντικός και μάλιστα γίνεται από χώρες έξω από την Ένωση, όπως δείχνει η χρηματοδότηση της Ρωσίας στις ε, διάφορες εξαρτήσεις όπως και ε, στη καταστροφή του Brexit που μόλις ανέφερε ο συνάδελφος. Οι γαλλικές εκλογές 2014 αυτά φαίνεται ότι επηρεάστηκαν. Επίση υπάρχουν υποψίες για ε, κινέζικη ε, παρακολούθηση. Αυτές οι απειλές δεν γνωρίζουν σύνορα. Μόνο μια κοινή ε, προσέγγιση της Ένωσης με κοινή προσπάθεια και θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ε, απειλές της Κίνας αλλά και τα ρωσικά τρόλ και θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπρέσο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξέτοιμοι συναδελφοί. Κυρία Επίτροπε. Η μαζική χρήση του ίντερνετ, η ψηφιοποίηση της οικονομίας μας, όπως πολλοί επεσήμαναν, δημιούργησαν μια νέα, ένα νέο στρατηγικό κίνδυνο και ανάγκη να εξασφαλίσουμε σε όλους τους πολίτες και ε, οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να ευημερούν σε προστατευμένους οικονομικούς ψηφιακούς χώρους σε μια χρονική στιγμή όπου συζητούμε για την ανάπτυξη του δικτύου 5G, των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει αλλά και των κινδύνων που μπορεί να κρύβει αλλά και τους κινδύνους ε, παρέμβαση της Ρωσίας και άλλων παραγόντων στις προσεχείς ευρωεκλογέ. Αυτό καθίσταται και μάλιστα μόλις ε, μερικές εβδομάδες πριν από τις ευρωπαϊκές ε, εκλογές. Αυτή η κίνδυνη είναι πολύ ορατή. Είδαμε και την Εστονία και την Γερμανία αντικείμενα συντονισμένων επιθέσεων. Πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση σε αυτούς τους κινδύνους. Η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει προτείνει κανονιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών είναι ευπρόσδεκτη, ωστόσο έχουμε καθυστερήσει σημαντικά. Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο Πρέπει να εξασφαλίσουμε περισσότερες επενδύσεις, να ενισχύσουμε το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, να αποφύγουμε παρεμβάσεις απαράδεκτες όπως αυτές ε, της Cambridge Analytica για, τις οποίες όλοι, για την οποία είμαστε όλοι ενημεροί. αυτό πρέπει να δράσουμε ταχύτατα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπρέσο. Ρουόνεν Λέρνεν, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σε ελεύθερε και ανώθευτε εκλογικέ αναμετρήσει, οι πολίτε εκφράζουν ελεύθερα την κατεύθυνση που θέλουν να λάβει η πολιτική στη χώρα τους. Στις επερχόμενες λοιπόν ευρωεκλογές τα αποτέλεσμα που θα βγει από την κάλπη έχει κρίσιμη σημασία λόγω και της μεταναστευτικής ε, κρίσης και του Brexit παρά αποκλίνουσες απόψεις που μπορεί να έχει ο καθένας μας. Συμφωνούμε οπωσδήποτε όλοι, είμαι βεβαία, πως πρέπει να προστατευτεί η δημοκρατία. Μόνο οι πολίτες πρέπει να είναι ε, σε θέση να αποφασίσουν την κατεύθυνση που θα λάβει η πολιτική ζωή στην Ευρώπη. Παρεμβάσεις από ξένα κράτη ή και με μονομένου άτομα, ε, με παραποίηση του αποτελέσματος των εκλογών, με διάδοση ε, παραπληροφόρηση ψευδών ειδήσεων, με hacking, με επιθέσεις σε εξυπηρετητές, πρέπει και να προβλεφθούν και να αποτραπούν εγκαίρως ε, δεν ε, είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να απαξιωθεί η εκλογική διαδικασία, να χάσει ο πολίτης την εμπιστοσύνη του στο αποτέλεσμα της κάλπης. Ε, σε μια περίοδο μάλιστα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά προσέλευσης της κάλπης για ορισμένα κράτη. Ευχαριστώ πολύ. Ζεκόφσκι, ένα λεπτό και 30 δεύτερα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ωραία συζήτηση. Καλή συζήτηση. Λέμε όλοι πως θέλουμε να κάνουμε περισσότερα ώστε να εξασφαλίσουμε πως οι επερχόμενες εκλογές θα είναι ανώθευτες ε, σε, μια, σε ένα περιβάλλον ε, κυβερνοασφάλειας θα διεξαχθούν. Αλλά να σας πω το εξή. Μήπως έρχεται όψιμα αυτή η συζήτηση. Ερχόμαστε εδώ να ανταλλάξουμε απόψεις ενώ θα έπρεπε να έχουμε αναλάβει δράση πολύ νωρίτερα εναντίον εκείνων των παραγόντων που έχουν και στο παρελθόν επηρεάσει την ετοιμιγωρία της κάλπης. Είμαι ευγνώμων για τις προτάσεις της Επιτροπής. Αλλά, κύριε Επιτροπέ, είμαστε και ειλικρινεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να προστατεύσουμε το, τον τρόπο διεξαγωγής των προσεχών ευρωεκλογών με το πακέτο αυτό. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά αυτή. Ακόμα και όταν δεν θα είστε πια επίτροπο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε πω στο μέλλον δεν θα υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστούν εκλογικέ αναμετρήσεις από οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα. Οι εκπρόσωποι όλων των πολιτικών ομάδων ε, είπαν ότι πρέπει να καταπολεμηθούν οι ψευδεί ειδήσει τα fake news, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί η ενημέρωση του πολίτη, πρέπει να εκπαιδευτεί ο πολίτης, να ξέρει πώς θα αναζητήσει την αλήθεια. Και έτσι απευθύνω έκκληση σε όλους σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ας στηρίξουμε τον πολίτη σε αυτή την αναζήτηση αλήθειας. Ο κύριος Μαριάς. Η ασφάλιση της αγκαιρεότητας των ευρωεκλογών είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να διασφαλίζουν την πολυφωνία. Όταν υπάρχει φήμωση και λογοκρισία, είναι βέβαιο ότι αυτό οδηγεί και σε fake news γιατί επί της ουσίας αποκρύπτεται η αλήθεια. έχω επανειλημμένα καταγγείλει εδώ τον αποκλεισμό και τη φήμωση του κινήματός μας ελλάδα ο άλλος δρόμος καθώς και τη δική μου φήμωση από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην ελλάδα είτε δημόσια είτε ιδιωτικά. δεν δίνουν την ευκαιρία προβολής των απόψεών μας. μας έχουν κυριολεκτικά φημώσει. ταυτόχρονα στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι δημοσκοπικές εταιρείες οι οποίες δεν βάζουν το κόμμα μας στο ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνουν στους πολίτες. με τέτοιους όρους δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία στην ελλάδα. δεν μπορούμε να πάμε σε ελεύθερες ευρωεκλογές στην ελλάδα και είναι κάτι το οποίο έχουμε καταγγείλει ως ecr και έχουμε στείλει και επιστολές διαμαρτυρίας και στα ίδια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις δημοσκοπικές εταιρείες και στον υπουργό εσωτερικών και θέλουμε κύριε επίτροπε την παρέμβασή σας. με τέτοιους όρους δεν διασφαλίζεται ελεύθερη κυκλοφορία ιδεών στις επερχόμενες ευρωεκλογές στην ελλάδα. κυριολεκτικά μας έχουν φημώσει. ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, Ω πρόεδρος τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, να πω λίγα λόγια για τη διάσταση εξωτερική πολιτική τη προστασία, τη ακαιρεότητα των επικείμενων ευρωεκλογών. Μόλι το Μάρτιο είχαμε τη δεύτερη έκθεση για την ε, στρατηγική επικοινωνική πολιτική για να αντιμετωπιστεί η προπαγάνδα από τρίτου εναντίον τη. Η έκθεση αυτή τόνισε πόσο ουσιώδη είναι η ελευθερία έκφραση και λόγου και η πολυφωνία των μέσων. Και εντοπίσαμε την ε, επιθετική καμπάνια της Μόσχας ως την κύρια πηγή παραπληροφόρησης. Γι' αυτό χαιρετίζω το ότι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αυξάνει την ε, αντίστοιχη task force για να είναι σε θέση να εντοπίζουν, να αναλύουν και να καταγγέλουν την παραπληροφόρηση. Συμφωνώ με πολλούς συναδέλφους που είπαν ότι επιπλέον πρέπει αυτά να γίνονται και σε επίπεδο κρατών μελών και σε νοσιακό επίπεδο. Να επερασπιστούμε τις ε, αξίες μας και τον κύβερνο πόλεμο μέσω ρωμαλαίων εκλογικών επικοινωνιών. Πρέπει να υπάρχει συνειδητοποίηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και των πλατφορμών δικτύωση. Και επιπλέον είναι ουσιώδε να βελτιωθεί ο τρόπο με τον οποίο εμεί ενημερώνουμε για τις αξίες μας και τις πολιτικές μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Μακάλιστερ, υπάρχει μια μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Υπάρχει ένα, μια μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Τη δέχεστε? Παρακαλώ κύριε Γκολνίσου. Ευχαριστώ αγαπητέ Αλφή Μακάλιστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μακάλιστερ, είπατε ότι οι ψευδείς ειδήσει προέρχονται από τη Μόσχα. Εγώ δεν θυμάμαι πολλά τέτοια παραδείγματα και ούτε είμαι εκπρόσωπος τύπου της ρωσικής κυβέρνησης. Αλλά ψεύτικες ειδήσει από τη Ρωσία παρόμοιες ε, έχετε με αυτές που ε, διασπείρει η Αμερικανική κυβέρνηση. Όταν ο Κόλλιν Πάουλ, για παράδειγμα, στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών είπε ότι έχει αποδείξεις για όπλα μαζικής καταστροφής, ενώ στην ουσία ήταν ε, τσιμέντο. Ευχαριστώ πολύ. Η απάντηση σας κύριε Μακάλιστα. Αγαπητέ συνάδελφε δεν ξέρω αν ε, θέλετε τώρα σοβαρή απάντηση στην ερώτησή σας. Ε, είναι σαφές ότι ένας εκπρόσωπος της άκρας δεξιάς στη Γαλλία δεν θα χάσει καμιά ευκαιρία να περασπιστεί το ρωσικό καθεστώ. Τον Μάρτιο, στην έκθεσή μα, είπαμε σαφώ. Υπάρχουν τεράστια έκταση προσπάθειε από πλευρά τη Ρωσία να υπονομευθεί η ευρωπαϊκή μα ενότητα. Και δεν είναι έκπληξη ότι ειδικά οι Ρώσοι στηρίζουν ενεργά κόμματα όπω το δικό σα. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που είστε αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που κάνετε έστω και απόπειρα να περασπιστείτε αυτέ τι δραστηριότητε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και τώρα... Διαδικασία κάτι στη Ο κύριο Κέλλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ε, ενδιαφέρουσα η συζήτηση ε, και, πολύ, και επικαιρή με έξι εβδομάδε να μένουν μόνο για τι ευρωεκλογέ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τι προτάσει και τι προσπάθειε για να βρει ε, λύσει για αυτή την πολύ ανησυχητική κατάσταση. σε προηγούμενη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο είπε πως ε, ε, τα περιστατικά παρέμβαση έχουν μειωθεί και βεβαίως θα πρέπει να ελπίζουμε θα μειωθούν περισσότερο. Απλώς ερωτώμες, ιδιαίτερα σε σχέση με όλες αυτές τις ψευδείς ε, ειδήσει και είμαι βέβαιος ότι αυτοί που θέλανε να ε, απειλούσαν μάλλον να δολοφονήσουν τον ε, φίλο μας ε, κύριο Τάραντ και αυτοί θα είχαν ψευδείς λογαριασμούς. Μήπως λοιπόν μπορούν να εντοπιστούν αυτοί οι ψευδείς λογαριασμοί πριν να γίνουν λογαριασμοί. Δηλαδή ξέρω εγώ να ζητούν το διαβατήριο για να μπορεί κανείς να αποδείξει την ταυτότητά του πριν φτιάξει λογαριασμό στο facebook ή τις άλλες προσχετικές πλατφόρμες. Γιατί διαφορετικά ατιμωρητή μπορεί κανείς να κάνει ό,τι θέλει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Ροζάτη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, Υπουργέ. Ε, είναι όντως ε, πολύ επικαιρό το θέμα. Όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, έχουμε όμως πολλές μαρτυρίες, πολλά σημάδια εχθρικής παρέμβαση σε διαφορετικές περιστάσεις στις ευρωπαϊκές εκλογές αλλά και εκτός Ευρώπης από τα ρωσικά τρόλ και που επηρεάζουν τους ε, ε, συμμετέχοντες στις εκλογές. Είναι κάτι που πρέπει πολύ σοβαρά να αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι μια πρακτική που υπονομεύει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε απλά να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια ε, ενώπιον τέτοιων πρακτικών. Θέλω να σας πω ότι πιστεύω πως η ανταλλαγή πληροφοριών, η ανταλλαγή ε, τέτοιων ε, πρακτικών, καλών πρακτικών δεν είναι σημαντική αλλά δεν είναι αρκή. Γιατί θα πρέπει νομίζω να αντιμετωπίσουμε αυτό, το, το, αυτές τις πρακτικές, να φτιάξουμε task force που να ασχολούνται μόνο με αυτό το ε, θέμα. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτήν την υπόθεση γιατί απειλεί την ενότητα και την ακυρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Λόπες Αγγιλιάρ. Κον ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Κίνγκ, η ελευθερία έκφραση δεν δίνει το δικαίωμα να προσβάλλει κανεί, να βρίζει ή να συκοφαντεί. Δεν δίνει το δικαίωμα να ψεύδεται, να χειραγωγεί. Ε, είναι όμω μια αρχική ε, και βασική αξία και η ανοιχτή κοινωνία είναι ευάλωτη και η δημοκρατία το ίδιο. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο πριν από, ε, μάλλον ενώπιον της ε, κυβερνοεπανάστασης η δημοκρατία να ε, εξοπλιστεί με μια διαδικασία κυβερνοασφάλειας για να καταπολεμήσει τα ψευδείς ειδήσει τις ε, ρητικές προπολέμους τρόλ και ψευδών ε, προφίλες στο διαδίκτυο. Ακριβώς έτσι ώστε να γίνεται μια συζήτηση όπως πρέπει πριν από τις ευρωεκλογέ. Όμως τίποτα από όλα αυτά δεν εμποδίζει τους ευρωπαϊστές να επικοινωνήσουν και να πούνε οι πρόκειται σε αυτέ τι ευρωεκλογέ. Πρόκειται για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ευρωπαϊκό δημοκρατικό χώρο με μια ανοιχτή συζήτηση, με μια κοινωνία που θα ενημερώνεται ελεύθερα. Είναι μια ευκαιρία ε, υπαρξιακής Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τόμασιτς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. είναι απαραίτητο να εμποδίσουν απόπειρε παρέμβαση στι ευρωπαϊκέ εκλογέ, αλλά και γενικότερα οι ευρωπαϊκέ δυνάμει πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ε, οι εκλογές να γίνουν με τρόπο αξιόπιστο και αυτό να επαληθευτεί με ε, ασφαλή κριτήρια και μέσα. Ωστόσο, δεν ε, μπορούμε να εξαντλήσουμε τις επικρίσεις μας στο να ρίχνουμε κατηγορίες κατά της Ρωσίας ή άλλων δυνάμεων. Μετά τις εκλογές θα, έχουμε πολύ φοβάμε θα έχουν πολύ φοβάμαι οι φεντεραλιστές μια μακρά περίοδο αντιμετώπισης της σκληρής αλήθειας, όπως άλλωστε συνέβη και στις Ηνωμένε πολιτείες. Πρόκειται για τις πολιτικές δυνάμεις που ηγήθηκαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί χρόνια, τις φεντεραλιστικές δυνάμεις που κανείς δεν θέλει. Ο πολίτης δεν θέλει μια, ενωμένη, μια Ευρώπη φεντεραλιστική και θα καταψηφίσει αυτές τις δυνάμεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί με προσέβαλα στο Twitter. Ένας πλαστός χρήστης και ένα πολιτικό κόμμα μου ζήτησε να το υποστηρίξω χωρίς να είμαι φίλος του στο Facebook. Σήμερα το πρωί κατάλαβα ότι πρέπει να έρθω σε αυτή τη συζήτηση. Όταν είδα ότι ήταν στη μέση διάταξη, και όχι για προσωπικού λόγου, γιατί αυτή η συζήτηση για τι επιθέσει κατά τη πολυφωνία, τι επιθέσει κατά τη δημοκρατία είναι ζωτική. Αυτό ο κυβερνοπόλεμο είναι πολύ πιο ευρύ από αυτήν την προσπάθεια τελευταία στιγμή. Πρέπει οπωσδήποτε να προλάβουμε του κινδύνου που σχετίζονται με την παραπληροφόρηση και τι ψευδεί ειδήσει. τα επεισόδια κυβερνοασφάλειας ε, στο facebook ε, δημοσιοποίησαν τα στοιχεία εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Είναι παρέμβαση και στην εκλογική διαδικασία. Αλλά πρέπει να ξέρουμε από ποιον γίνεται. Γίνονται από τα κόμματα της ακροδεξιάς. Είναι τα κόμματα που καλούν στην ξενοφοβία, το μίσος και που έχουν ένα λόγο ρατσιστικό και ξενοφοβικό. Το βλέπουμε και στην Ισπανία αυτό. Η κατάργηση των πλαστών χρηστών του Twitter και του Facebook είναι υποχρέωση. Πρέπει αυτά να ελέγχονται και ε, εκτός ε, ίντερνετ. Πρέπει να υπάρχει πολιτική διαφάνεια. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γραπίνη. Α, έχει φύγει. Ζολογεύσκη. Τελευταίος. Πρόεδρε, επί δύο χρόνια ε, συμμετείχα σε εργασίες της Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, όπου συζητήθηκε επανειλημμένο το θέμα της ε, κυβερνοεγκληματικότητας και της κυβερνοάμυνας. Οι πληροφορίες που λάβαμε και θέλω να το τονίσω αυτό για τρομοκράτες ε, που δρούσαν όχι μόνο μέσω τοποθέτησης μιας βόμβας αλλά και μέσω εκρηκτικών ε, ψευδών ειδήσεων και υπονόμευσης της ε, πραγματικότητας ε, είναι πολύ σημαντικές. Μιλήσαμε βέβαια και για τους πληροφοριοδότες, τους whistleblowers και πρέπει να τους προστατέψουμε. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτούς και εκείνους που επαληθεύουν τις ειδήσει και μπορούν να διαδώσουν ασφαλείς πληροφορίες για την για τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργάνων, ταυτόχρονα πρέπει να καταπολεμήσουμε όλους εκείνους οι οποίοι κατασκευάζουν ψευδείς ειδήσει, ψευδή μηνύματα ψευτοκατηγορίες κατά των πολιτικών κομμάτων ή και των ιδιωτών στην Ευρώπη. Για να είναι ασφαλής η Ευρώπη πρέπει να είναι ασφαλές και το σύστημα ενημέρωσης. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ο πολίτης να έχει την αίσθηση ότι εάν υπάρχει κάποια τέτοια ε, εγκληματική δραστηριότητα θα παταχθεί. Και έτσι μπορούμε να αποκαταστήσουμε τους ε, την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ για να απαντήσει ο εκ μέρους Ευρωπαϊκή Επιτροπής, ο Επίτροπο Κίνγκ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τη συζήτηση. Θα ήθελα να τοποθετηθώ σε δύο μόνο σημεία. Πρώτα απ' όλα από βουλευτές που βρίσκονται πίσω ε, από τη θέση στην οποία κάθομαι εγώ ακούστηκε ότι αυτό που κάνουμε ισοδυναμεί με φήμωση του ελεύθερου λόγου ότι είναι δηλαδή λογοκρισία. Θέλω να είμαι απολύτω σαφής ότι ποτέ δεν υπενηχθήκαμε, ούτε και πρόκειται ποτέ να υπενηχθούμε ότι κάποιος είτε πρόκειται για δημόσια αρχή, για αρχή ή ακόμα λιγότερο για ιδιωτικό φορέα, έχει την ευθύνη να επαληθεύσει εάν είναι σωστή, ακριβής, ψευδής, λάθος ή κακιά, κακή μία πληροφορία. Εδώ θέλουμε να έχουμε μέτρα προαγωγής περισσότερης διαφάνειας που θα ε, πλαισιώνει τον πολιτικό διάλογο περισσότερης διαφάνειας για το προέλευση των πληροφοριών από πού βγήκαν, από πού προέρχονται ώστε εμείς ως πολίτες να μπορούμε καλύτερα να αξιολογούμε τις πληροφορίες αυτές και να διαμορφώνουμε γνώμη. Αυτό σημαίνουν τα μέτρα τα οποία μέσω του κώδικα προάγουμε περισσότερη δηλαδή διαφάνεια σε σχέση με την πολιτική διαφήμιση, το περιεχόμενο χορηγίας, την ανάπτυξη και δημιουργία νέων λογαριασμών, επαλήθευση γεγονότων που μεταδίδονται μέσω των ειδήσεων, να επαληθεύεται λοιπόν ώστε να ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα από αυτές τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, εάν υπάρχει αποδεδειγμένα δε παραπληροφόρηση, να γίνεται και η σχετική αποκατάσταση της αλήθειας. Αυτή είναι για μένα η ουσία της προάσπισης του ελεύθερου λόγου, Ελευθερία ενημέρωσης και πόρο απέχει από οποιαδήποτε έννοια λογοκρισίας. Δεύτερη παρατήρηση και αντίδραση σε επισημάνσεις, η σημασία της ανθεκτικότητάς μας στις κυβερνοεπιθέσεις. Η παρέμβαση μέσω του κυβερνοχώρου είναι ε, στοιχείο άκρος ουσιώδες και απαραίτητο και γι' αυτό το νομοθέτημα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που υιοθετήσατε εσείς ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία όπως και η σχετική υπηρεσία. Πολύ όμως υπογραμμίσατε ότι πρέπει και να προχωρήσει σε υλοποίηση το νομοθέτημα αυτό. Σας βεβαιώ λοιπόν από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για ουσιαστική υλοποίηση του νομοθετήματος για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ελπίζω επί τη ευκαιρία ότι θα στηρίξετε και τα κέντρα ε, δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας που θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της ανθεκτικότητας, της κυβερνοανθεκτικότητάς μας. Θα έχουμε να κάνουμε λοιπόν με τον σχεδιασμό ενός σκελετού της συζήτησης για τα μέτρα στον κυβερνοχώρο. Γι' αυτό έχουμε τώρα τα μέτρα επαλήθευσης, γι' αυτό έχουμε τα μέτρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ώστε να αντιληφθεί ο πολίτης τη σημασία όχι μόνο της ε, ψηφιακής ε, ασφάλειας σε όρους κόστους, τιμήματος ή τιμής, αλλά και την ε, διάσταση της ασφάλειας σε όλα αυτά. Ο Αβραάμ Λινκόλν είχε πει ότι οι εκλογές ε, ανήκουν στο λαό και την απόφαση τη λαμβάνει ο λαός μέσω των εκλογών. αυτό πρέπει και εμείς να υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η Υπουργός κ. Τσότα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ε, κύριοι Ευρωβουλευτές, ε, Κύριε Επίτροπε, είναι καθήκον μας να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως η ελευθερία λόγου, το, η ελευθεροτυπία και η ελευθερία του ε, συνεταιρίζεσαι. Δεν μπορούμε να είμαστε ε, ε, οι Αυτές οι εκλογές δεν θα είναι όπως ε, συνηθίζεται και οι πολίτες μας έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν ελεύθερα. Πρέπει να υπερασπιστούμε τις ευρωπαϊκές αρχές. Τα ευρωπαϊκά όργανα και κράτη-μέλη δεν εφίστησαν προσπαθειών για να εξασφαλίσουν την τήρηση αυτών των αρχών. Προσπαθούμε να μάθουμε από αλλήλους μέσω της μοιρασίας των καλύτερων πρακτικών. Επίση, ε, θεσπίζουμε μέτρα που ενθαρρύνουν την περισσότερη επιγραμμική ασφάλεια, την λογοδοσία και την κεραιότητα. Ε, εξασφαλίζουμε με τον κανονισμό προστασία των, ε, των δεδομένων και προστασία των ηλεκτρολογικών συστημάτων και υποδομών. Επίση είναι κρίσιμη η ανθεκτικότητα ε, των συστημάτων μας. Θα παραθέσω από το, ε, από το 1984 τον George Orwell ε, που, έλεγε ότι η εξουσία είναι αυτή που κατακαιρματίζει το ανθρώπινο μυαλό σε κομμάτια τα οποία μετά ξανασυναρμολογεί όπως επιθυμεί. κάποιοι θέλουν έτσι να συναρμολογήσουν το εγκεφάλους των ψηφοφόρων μας δίνοντάς τους συγκεκριμένες πληροφορίες ή ψευδείς ειδήσει. Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τους συμπολίτε μας από αυτές τις δυνάμεις. Το οφείλουμε στους συμπολίτε μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Υπουργέ, ευχαριστώ Επίτροπε που ήσασταν σήμερα εδώ. Η κοινή συζήτηση ολοκληρώνεται εδώ. Χθε ο πρόεδρο ανήγγειλε δύο ερμηνείε του κανονισμού που προτάθηκε από την Επιτροπή, προτάθηκαν από την Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων. Η ομάδα EFTD υπέβαλε μία ένσταση στην ερμηνεία του άρθρου 32, πέμπτη παράγραφος, πρώτη υποπαράγραφος, δεύτερο εδάφιο. Αυτή η ερμηνεία αυτού του άρθρου θα ψηφιστεί αύριο. Όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 149α, δεύτερη παράγραφος, δεν υπευλήθησαν ενστάσεις εντός της προθεσμίας των 24 ωρών. Αυτή η ερμηνεία λοιπόν θεωρεί, θεωρείται ότι ενεκρίθη σύμφωνα με το άρθρο 226. Σε σχέση με την κοινή θέση για την επέκταση του καταπεστα... καταπιστεύματος της Ένωσης για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που εστάλει στον πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης και στην Επιτροπή Προπολογισμών, όπω αναγγέλθη χθε στην έναρξη τη συνεδρίαση, δεν υπερβήθησαν αντιρρήσει εντό τη προθεσμία των 24 ωρών. Ο πρόεδρο λοιπόν θα αποστείλει επισήμω αυτή την κοινή θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα έχουμε την κοινή συζήτηση που αφορά τον ορίζοντα Ευρώπη έκθεση του κυρίου Νίκα και του κυρίου Έλερ και δίνω το λόγο στον εισηγητή κύριο Νίκα για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε αγαπητή αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρετε. Τέσσερις μήνες μετά την συζήτηση στην Ολομέλεια πριν από τις συνομιλίες και δέκα μήνες αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε το πρόγραμμα πλαίσιο για την καινοτομία και την έρευνα ορίζων Ευρώπη, να είμαστε πάλι εδώ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό για το μέλλον, ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να επηρεάσει το μέλλον, την έρευνα, την ανάπτυξη, την οικονομία και το επίπεδο διαβίωσης στην Ευρώπη με την ε, επιστήμη, την καινοτομία ε, μπορεί η Ευρώπη να καταστεί ανταγωνιστική, να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στο διεθνές επίπεδο και να δημιουργήσει ποιοτικέ θέσεις εργασίας. Μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω πως οι συνομιλίες των οποίων ηγήθηκα στέφθηκαν με μερική επιτυχία και να σας εξηγήσω γιατί. Η αρχή της αριστείας διατηρείται στην επιλογή των προγραμμάτων ένα 30% των προϋπολογισμών θα αξιοποιείται για την υλοποίηση των στόχων του τοί κλιματικής αλλαγής, δηλαδή θα γίνεται επιλογή ε, προγραμμάτων με περιβαλλοντικό χαρακτήρα και προσθέμενη αξία για το υλικό χρήστη. Επίσης, τα μέσα μικρομεσαίων επιχειρήσεων διατηρούνται με, σε μορφή αντίστοιχη με αυτή που είχαμε στο τελευταίο το 2000 και με ένα ποσοστό 20% ε, χορηγίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προβλέπεται όπως και στο παρελθόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η απόκληση μεταξύ έρευνας και καινοτομίας μειώνεται γιατί θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 3,3% στο πρόγραμμα πλαίσιο κράτη τα οποία ε, υστερούν και αυτό οφείλεται σε μία ρήτρα που ονομάζεται widening του προγράμματος. Έτσι λοιπόν μπορεί η Ευρώπη να προχωρήσει πιο ομοιόμορφα και συνεκτικά στην έρευνα και την καινοτομία. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας συνεχίζει τις εργασίες του, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, εξασφαλίζει αυτά αποτελέσματα για όλους τους Ευρωπαίους, πέντε τομείς, πέντε ε, εντολές ορίζονται όπως η κλιματική αλλαγή, ο καρκίνος, η καθαρή ωκεανή, η αντιμετώπιση των κλιματικών προβλημάτων, η διατροφή και το έδαφος, τα εδάφη και πρέπει να γίνει τώρα πια η επιλογή των πρώτων αποστολών που θα αντιστοιχούν στα κριτήρια αυτά. Έχουμε τώρα δώσει μεγάλη έμφαση με τα πρώτα προγράμματα ορίζον, ε, του ορίζοντα ε, στην καινοτομία. Πρέπει πλέον να δώσουμε έμφαση εξίσου και στην έρευνα και μάλιστα στην έρευνα βάση, στη θεμελιώδη έρευνα, η οποία είναι εκ των κάνε φόρος για την ε, ανταπόκριση που θα δώσουμε στους στόχους του προγράμματος. Και αυτό βεβαίως θα πρέπει να συνοδευτεί από μια απλούστευση, από λιγότερο γραφειοκρατικό άχθος και διευκόλυνση των ε, εταίρων. Το Κοινοβούλιο έδειξε ιδιαίτερα, ε, ιδιαίτερη ευμένεια και εξυπηρέτησε στενά ε, χρονοδιαγράμματα προκειμένου να προχωρήσει η συμφωνία έστω και μερική στην ψηφοφορία αύριο, αποδεικνύοντας έτσι την προσήλωσή του στην εξυπηρέτηση συμφέροντος των πολιτών και των αναγκών των επιστημόνων. Υπάρχουν ζητήματα που δεν συζητήθηκαν, ο προπολογισμό για τις διεθνείς σχέσεις και συνεργασία. Ωστόσο, δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε επίπεδο υψηλό φιλοδοξιών και εν ώψη του προσεχούς κοινοβουλίου με 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι η σε περίοδος θα έχει πολύ καλή πολύ καλή χρηματοδότηση. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την πολύ καλή υποστήριξη που μας προσέφερε. Είναι καλά τα αποτελέσματα και ευχαριστώ τους συναδέλφους που δεν είναι όλοι εδώ, λίγοι μάλλον είναι παρόντες. Πάντως είχαμε πολύ καλή συνεργασία και μπορούμε να υπερηφανευόμαστε για μία πρώτη ομόφωνη απόφαση με υποστήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες. Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα με το Horizon 2020. Ε, Κύριος Χέλλερ, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Καλημέρα νομίζω είναι σήμερα για την Ευρώπη. Και καλύτερα αύριο που θα ψηφίσουμε το πρόγραμμα. Η Ευρώπη έχει φιλοδοξίες. Αύριο θα αποκτήσουμε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα μη στρατιωτικής ε, πολιτικής έρευνας στον κόσμο. Και το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται προς τους πολίτες της Ευρώπης. Συζητάμε αυτές τις μέρες για την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας για την ε, κλιματική αλλαγή. 35% της έρευνας στην Ευρώπη θα ασχοληθεί με την κλιματική αλλαγή. Επίσης η υγεία των συμπολιτών μας μας απασχολεί. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τον καρκίνο. Θέλει, ιδιαίτερα τον, καρκίνο, τον παιδικό καρκίνο. Και μας ενδιαφέρει και η ασφάλεια των τροφίμων. Και η πολιτιστική μας κληρονομιά. Με νέους ε, τομείς όπως ε, ο ψηφιακός τομέας και ο δημιουργικός κλάδος. Είναι λοιπόν φιλόδοξο αυτό το πρόγραμμα. Είναι φιλόδοξο με παγκόσμια κριτήρια. Το πρόγραμμα για την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα. Οι φιλοδοξίε μα για τι νέε ξεβαντικέ τεχνολογίε. Το θέμα τη ψηφιοποίηση των διαδικασιών παραγωγής στην Ευρώπη. Αυτή είναι τομεί μέλλοντος, τομεί εχμή για την ευρωπαϊκή έρευνα θα βοηθήσουν και την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και τους συμπολίτες μας. Εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, την υγεία τους, τα πιο άμεσα αιτήματά τους. Δεν είναι θεωρητική αφηρημένη συζήτηση για την πολιτική έρευνα. Είναι η βάση για την Ευρώπη. Ζούμε σε μια Ευρώπη υψηλών αποδοχών. Σε μια Ήπειρο όπου έχουμε το υψηλότερο επίπεδο κοινωνικών δαπανών στον κόσμο. Και ο λόγος που είμαστε ανταγωνιστική παρόλα αυτά είναι η καινοτομία και η έρευνα. Από το 18ο αιώνα ήταν η Ευρώπη ο χώρος όπου έγινε περισσότερη καινοτομία, κοινωνική ανάπτυξη, έρευνα. Είναι η βάση επί της οποίας δημιουργήσαμε τη σημερινή Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, η συνολική κοινωνική ευθύνη για την ελευθερία, την ασφάλεια, για τη δημοκρατία, αλλά και για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, όπως κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά βρίσκουν τη θέση τους σε αυτό το πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστικοί. Σε τι κόσμο βρισκόμαστε με αυτό το πρόγραμμα που απαιτεί 120 δις για αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κινούμεθα σε ένα κόσμο ο οποίος αλλάζει με φρενήρη ρυθμό. Και μεταξύ των 10 μεγαλύτερων ερευνητικών επιχειρήσεων στον κόσμο, των 10 επιχειρήσεων που κάνουν την περισσότερη έρευνα, είναι μόνο μία ευρωπαϊκή. Και μεταξύ των 20 μεγαλύτερων μόνο τρει Από αυτέ τις τρει επιχειρήσεις, οι δύο είναι αυτοκινητοβιομηχανίε. Η Amazon, για παράδειγμα, το 2017 δαπάνησε 20 δισεκατομμύρια δολάρια για την έρευνα. Είναι περισσότερα από ό,τι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπάνησε για την έρευνα το 2017 ακριβώς. Το πρόγραμμα αυτό και νομίζω είναι ένα σημαντικό βήμα για να επανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας αλλά και για να έχουμε την κυριαρχία στον τομέα αυτό στην Ευρώπη. Αυτές τις μέρες συζητάμε για κλιματική αλλαγή αλλά πρέπει να δούμε και εμείς. Κάνουμε αρκετά γι' αυτό. Είμαστε αρκετά φιλόδοξοι. Πώς συμβάλλουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε αρκετά υπερήφανοι για να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα έρευνα εγγυάται ότι θα υπάρχει τουλάχιστον έρευνα για την ε, κλιματική αλλαγή. Στην ε, Αμερική μειώθηκαν οι πόροι. Απολύθηκαν 3.000 υπάλληλοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντο. Η Κίνα δεν είναι καθόλου φιλόδοξη σε αυτό το τομέα. Η Ευρώπη όμω έχει αποτελέσματα. Αυτό το πρόγραμμα έρευνα θα έχει αποφασιστική σημασία και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Είχαμε ταχύτατα αποτελέσματα, ιστορικά μικρό το χρονικό διάστημα. Υπάρχει ασφάλεια για αυτού που θα εμπλακούν και καταδείξαμε ότι μπορεί γρήγορα και αποτελεσματικά να δράσει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ο κύριο Μοέντας, παρακαλούμε εκ μέρους της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Την τελευταία φορά που είχα την τιμή να απευθυνθώ σε αυτή την Ολομέλεια ήταν η 11η Δεκεμβρίου πέρυσι και τότε καλωσόρισα την πολιτική συνένεση η οποία προέκυψε στην Επιτροπή Ήτρε και ευχαριστώ τον Πρόεδρο Μπούζεκ την ικανότητα, για την ικανότητά σας ε, να δουλέψετε ποιοτικά και γρήγορα. Αυτή ήταν η φιλοδοξία του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον κρονισμό πλαίσιο που θεσπίζει τον ορίζοντα Ευρώπη και τις σχετικές προτάσεις ε, για το πρόγραμμα. Ανοίγει το δρόμο για το Συμβούλιο και για την Επιτροπή ώστε να διαπραγματευτούν πραγματικά. Και να είμαστε ξανά μετά από τέσσερις μήνες και έξι τριμερείς ε, διαλόγους και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε επιτύχει μια τόσο ισορροπή συμφωνία όσον αφορά τον οριζόντα Ευρώπη. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια κύριε Νίκα, συγχαρητήρια κύριε Έλερ για την καταπληκτική δουλειά που κάνατε. Έχω εντυπωσιαστεί. Εντυπωσιαστικά πώς τα καταφέρατε, πώς επιτύχατε μια συνένεση, πώς εργαστήκατε τόσο σκληρά, πώς όλοι εργάστηκαν τόσο σκληρά. Τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια λοιπόν. Θα παρακολουθώ αύριο για την επιβεβαίωση, την επικύρωση. Θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο Μπούζεκ που πάντα ήταν εκεί στην Επιτροπή Ήτρε και ή μαζί μας και συγχαρητήρια και στο Συμβούλιο. Συγχαρητήρια στη Ρουμανική Προεδρία και θα ήθελα τώρα να μιλήσω λίγο προσωπικά. Συγχαρητήρια κύριε Πρέσβη, σε εσά και στην ομάδα σα. Εργαστήκατε πολύ σκληρά, 24 ώρε το 24ωρο, για να επιτύχετε όλα αυτά. Και σα είμαι ευγνώμων. Last week. Την περασμένη εβδομάδα ζήσαμε μια όμορφη στιγμή. Νομίζω ότι ζήσαμε όλοι αυτή την όμορφη στιγμή όπου για πρώτη φορά στη ζωή μας είδαμε μία φωτογραφία μιας μαύρης τρύπας. Φανταστείτε, πριν από 100 χρόνια ο Αλβέρτος Άινστάιν φαντάστηκε μία μαύρη τρύπα και για 100 χρόνια οι άνθρωποι προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι είχε δίκιο. Και τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε και η Ευρώπη ήταν παρούσα. Πάτησε το κομπάκι που έδειξε αυτή την εικόνα αυτή τη φωτογραφία που έδωσε στον κόσμο πράγματα που δεν είχε φανταστεί ποτέ διότι ο Αϊνστάιν ούτε αυτός δεν μπορούσε να φανταστεί τι είχε πετύχει, πόσο αυτό θα είχε επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο. Υπήρξε ένας επιστήμονας που είπε ότι, ξέρετε, η επιστήμη είχε ιστορία πριν από αυτή τη στιγμή, πριν τη φωτογραφία και μετά θα έχουμε μια νέα ιστορία μετά από αυτή τη χρονική στιγμή. Νομίζω ότι αυτό για μένα θα ήταν η στιγμή που περιγράφει ολόκληρη την ευρωπαϊκή επιστήμη. Είναι η στιγμή που περιγράφει ε, την ανοιχτή επιστήμη, την ανοιχτή καινοτομία, το άνοιγμα προς ολόκληρο τον κόσμο. Διότι σε εκείνη την αίθουσα, εκείνη την ημέρα, εκπροσωπούσαν 200 επιστήμονες, 40 διαφορετικές εθνικότητες. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα περήφανος διότι ορίζοντας Ευρώπη αφορά ακριβώς αυτό την πρωτοπορία μας ε, στις επιστήμες ως ε, Ευρωπαίων. Αν σκεφτείτε τι έχουμε επιτύχει, ε, τι αποφασίσαμε για το επόμενο πρόγραμμα, όλες αυτές τις αποστολές, όπως αναφέρθηκε ο κ. Σέλλα, επιστημονικές αποστολές που θα είναι κατανοητές στους ανθρώπους, που θα κοινοποιούμε στους ανθρώπους για τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε για να θεραπεύσουμε ασθένειες όπως το καρκίνο. Αυτό θα μας συνδέσει με τους λαούς μας και οι προσπάθειε που θα κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η καινοτομία όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση τη καινοτομία, οι εταιρικέ σχέσει που αποφασίσαμε να επιλέξουμε για ευ... και ευκολότερος τρόπος καθορισμού αυτών των εταιρικών σχέσεων και κάτι πολύ σημαντικό για όλου μα. Το πρόγραμμα αφορά την αριστεία. Πρέπει όμω να βοηθήσουμε και εκείνου που ε, φιλοδοξούν να επιτύχουν την αριστεία. Και αυτό το χρωστάμε σε εσά, στο Κοινοβούλιο. Το ότι επιτύχαμε αυτή τη συμφωνία, το ότι θα αφιερώσουμε 3,3% του προπολογισμού για ε, τη διεύρυνση των μέτρων στο μέλλον.